Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Δεν έχουμε μόνιμο εισηγητή, γιατί θα οριστεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Τρόικα των αποκεντρωμένων οργανισμών. Είναι η αιτήσια συνεδρίασή μας. Τη απουσία λοιπόν του μόνιμου εισηγητή θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Σιλβάνο Πρέσα που είναι ε, διευθυντής ε, της Γενικής Διεύθυνσης Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας εξηγήσει ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για το 2015. Θα μας μιλήσει επίσης και για την γενικότερη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της μείωσης του προσωπικού μέχρι τα τέλη του 2017. Γιατί αυτή είναι η γενική τάση. Είναι αυτό που περιμένουμε να γίνει για να μειωθούν οι δαπάνες. Αφού ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σιλβάνο Πρέσα, μετά θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τον κύριο Μόρτον Κέρουμ, ο οποίος εκπροσωπεί τους οργανισμούς. Εκείνος θα εκφράσει τη δικιά τους άποψη για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεχομένως θα ακούσουμε και τη θέση της Κορεπέρ της προηγούμενης εβδομάδας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε μπροστά σας ένα λεπτομερές έγγραφο το οποίο προετοιμάστηκε από τους ίδιους τους οργανισμούς και έχει διανεμηθεί τα μέλη της Επιτροπής μας ήδη από το πρωί. Κύριε Σιλβάνο Πρέσα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας πω δύο λόγια για τη διαδρομή πρώτα απ' όλα των αποκεντρωμένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ασχοληθώ κυρίως με την κατάσταση πραγμάτων σήμερα. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Έλεγα λοιπόν ότι τα τελευταία 35 χρόνια 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί δημιουργήθηκαν με διάφορα καθήκοντα, ποικίλα. Η αύξηση αυτή βέβαια έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε και αντικατοπτρίζεται στα ποσά στη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προπολογισμό, η οποία αυξήθηκε από το 2000 εννέα φορές και τώρα είναι πάνω από 800 εκατομμύρια ετησίως το κόστος των κοινοτικών προπολογισμό. Το ίδιο βλέπουμε και όσον αφορά το συνολικό προσωπικό, τις θέσεις δηλαδή που προβλέπονται για τους οργανισμούς. Έχουν αυξηθεί πάνω από τέσσερις φορές από το 2000 μέχρι τώρα. Και είναι πάνω από 6.000 στις, στους 32 αυτούς οργανισμούς. Υπήρξε λοιπόν μεγάλη ανάπτυξη στους οργανισμούς. Τώρα το πλαίσιο ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια είναι ένα πλαίσιο μάλλον παγίωσης όσον αφορά τον κοινοτικό προπολογισμό και πρόκειται επίση και για μια απαγίωση και όσον αφορά τα θεσμικά όργανα αλλά και τους απαγκεντρωμένους αυτούς οργανισμούς. Αυτό φαίνεται και στην Διοργανική Συμφωνία. Εκεί βλέπουμε κάποια στοιχεία από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Εκεί αναφέρεται πολύ συγκεκριμένο στόχος που είναι η μείωση κατά 5% τον ε, αριθμό των θέσεων, του προσωπικού δηλαδή, σε όλα τα όργανα και όλους τους οργανισμούς μέσα σε πέντε χρόνια. Στην περίπτωση των αποκεντρωμένων οργανισμών, οι προσπάθειες αυτές γίνονται πιο περίπλοκες επειδή δεν είναι ε, εντελώ ε, έτοιμοι όλοι οι οργανισμοί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι παλιότεροι βέβαια, έχουν εγκαθιδρυθεί πλήρω, αλλά υπάρχει μια άλλη ομάδα οργανισμών που δημιουργήθηκαν πιο πρόσφατα και που ακόμα δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο κανονικής λειτουργίας ώστε να φέρουν πλήρως πέρας τα καθήκοντά τους. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία οργανισμών, που είναι βέβαια πιο παλιοί οργανισμοί και που ο στόχος τους, τα καθήκοντά τους έχουν πρόσφατα επεκταθεί. Αυτό σημαίνει ότι στον προγραμματισμό και στην ομοθετική διαδικασία που τους δημιούργησε ή που επέκτηνε τις αρμοδιότητές τους, των οργανισμών αυτών, εκεί βλέπουμε ότι χρειάζονται και επιπλέον πόροι και επιπλέον προσωπικό. Οπότε υπάρχει εδώ μια εκτίμηση για 300 επιπλέον θέσεις που πρέπει να προσθεθούν στην σημερινή δομή. Όταν βλέπουμε λοιπόν τους στόχους που υπάρχουν στη Διοργανική Συμφωνία, υπάρχει ο γενικός στόχος της μείωσης του 5% του προσωπικού, αυτό σημαίνει 300 θέσεις λιγότερο για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς συνολικά. Βλέπουμε όμως και μια αύξηση κατά 300 προκειμένου να φέρουν σε πέρα στα νέα καθήκοντα και να επιτρέψουν στους πιο πρόσφατους οργανισμούς να φτάσουν σε ένα κανονικό επίπεδο εργασίας. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό, εφόσον φαίνεται παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να το πετύχει αυτό με ανακοίνωση η οποία παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2013. Προκειμένου λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα αύξησης του προσωπικού σε ορισμένους οργανισμούς μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της μείωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πουλ με κάποιο είδου μόχλευση για τους ε, οργανισμούς εκείνους οι οποίοι φτάνουν στον κανονικό ρυθμό λειτουργίας τους και αρχίζουν να σταθεροποιούνται. Με 1% δηλαδή το χρόνο. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα σύνολο θέσεων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθηθούν οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν επιπλέον καθήκοντα από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Ο ρυθμός βέβαια της μείωσης και της αύξησης πρέπει να καταλήξει σε κάποια ισορροπία. Η δυνατότητα και η ταχύτητα, δηλαδή για να δημιουργηθεί αυτό το πουλ, καθορίζει πόσο γρήγορα μπορούν να ενισχυθούν και οι οργανισμοί που έχουν ανάγκη από ενίσχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έκανε μία πρόταση για προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων όλων των αποκεντρωμένων οργανισμών και των τριών κατηγοριών, κοιτώντα τον κάθε οργανισμό χωριστά και εκτιμώντα τι ανάγκε που υπάρχουν σε αυτού των οποίων τα καθήκοντα επεκτάθηκαν ή που είναι πιο νέοι. Και αυτά μέχρι το 2020. Στη μείωση τώρα πέρα από το 5% για τους οργανισμούς που φτάνουν σε κανονική πορεία, σημαίνει ότι πρέπει να δούμε και τους υπόλοιπους οργανισμούς, πώς και αυτοί φέρνουν σε πέρα τα καθήκοντά τους. Ο προγραμματισμός λοιπόν των ανθρώπινων πόρων φαίνεται και από την συνεισφορά από τον προπολογισμό στον κάθε οργανισμό. Θέλουμε βέβαια όλα αυτά να είναι συμβατά με, τα, με τις υποοροφές τις οποίες καταλήξαμε με τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 14 20. Η κάθε οροφή για δαπάνες έχει και υποοροφές ενδεικτικές ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι δαπάνες θα ανταποκρίνονται απόλυτα στις οροφές και ότι το σύνολο των δαπανών θα παραμένει στα επίπεδα οροφής δαπανών όπως αποφασίστηκαν. Ο προγραμματισμός λοιπόν που ε, προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα 7 χρόνια ε, σέβεται το ανώτατο αυτό επίπεδο και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει και απόλυτη συνοχή με τον στόχο που μιλάει για μείωση κατά 5% του προσωπικού σε συνολικά σε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και προβλέπει μάλιστα και ένα πλαίσιο πρόβλεψης για τους οργανισμούς και για την προετοιμασία του ετήσιου προπολογισμού. Και μάλιστα για πρώτη φορά έγινε αυτό για το 2014, όπου το συνολικό, ο συνολικός αριθμός θέσεων σε όλους τους οργανισμούς μειώθηκε λίγο μετά τις διαπραγματεύσεις, αλλά μειώθηκε. Άρα εδώ οι προσπάθειες αυτές μείωσης του προσωπικού είναι πραγματικές, το βλέπουμε. Τώρα έρχομαι στο σχέδιο προπολογισμού για το 2015. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της ακολούθησε τον Γενικό Προγραμματισμό Ανθρωπίνων Πόρων με τα ποσά που δίνονται συνολικά ή εν μέρη από τον κοινοτικό προπολογισμό για τους οργανισμούς αυτούς, λαμβάνοντα υπόψη τις ανάγκες έτσι όπως έχουν εκτιμηθεί. Οι αποφάσεις τώρα που λήφθησαν από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο για το 2014 λαμβάνονται επίσης υπόψη, γι' αυτό και δίνονται κάποιες επιπλέον θέσεις σε ορισμένους οργανισμούς. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο για το γενικό πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα χρόνο. Και αυτό είναι ότι υπάρχει ένα νέο σώμα το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο ονομάζεται Single Resolution Board για τον τραπεζικό τομέα. Πρόκειται για ένα νέο σώμα για το οποίο 122 θέσεις επιπλέον θα δημιουργηθούν το 2015. Πρόκειται για αρχική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και σήμερα το πρωί η Επιτροπή σας ενέκρινε μια προσωρινή μεταφορά για να αρχίσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά από το 2015 το νέο αυτό σώμα, το νέο Συμβούλιο Εξυγίανση δηλαδή, θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρω και θα επιστρέψει στον προπολογισμό την προκαταβολή. Λίγο πολύ εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Κάτι σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σίγουρα το γνωρίζετε περισσότεροι από εσά είναι η δημιουργία μιας διοργανικής ομάδας εργασίας. Μια τέτοια διοργανική ομάδα εργασίας συμφωνήθηκε στα πλαίσια του προπολογισμού 2014. Την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλιστα. Δύο φορές έχει συνεδριάσει η ομάδα αυτή, έχει αποφασιστεί η σύνθεση, η μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα. Και όσον αφορά την εντολή, η ομάδα αυτή εργασίας θα προσπαθήσει να βρει τρόπους για να καθορίσει πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντα των οργανισμών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου να μειωθεί το προσωπικό τους κατά 5% όπως συμφωνήθηκε στη Διοργανική Συμφωνία. Δεύτερον, θα εξετάσει τρόπους για να επιτεθούν συνεργίες προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλη με διαφορετικό όμως τρόπο υπέρ της μείωσης αυτής του προσωπικού. Και τρίτον θα προσπαθήσει να βρει τρόπους για κατάλληλες υποχρεώσεις και προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθούν οι οργανισμοί σε επιπλέον καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει νομοθετικές αρχές. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την προσέγγιση ακολούθησε για να καταλήξει στην πρότασή της όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τον προπολογισμό τους για το έτος 2015. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, αφού ακούσαμε τη θέση της Κομισιόν για το δημοσιονομικό πλαίσιο των οργανισμών, και την ανάγκη μείωσης του προσωπικού, αντιμετωπίζοντας ωστόσο τη δημιουργία νέων οργανισμών, νέων δομών και το πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία, θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Μόρτιν Γερούμ, που είναι ο εκπρόσωπος των οργανισμών, να μας δώσει τη δική του αξιολόγηση. Very much, Mr. Chairman. Vice Chairs, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδροι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2015. Καταρχήν είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας συγχαρώ για την ε, εκλογή σας εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Οργανισμών τους οποίους αντιπροσωπεύω σήμερα εδώ. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι προσβλέπουμε πολύ στη συνεργασία μαζί σας τα επόμενα χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως είμαστε πως έχουμε ένα ήδη υπάρχουν θεμέλιο, την συνεργασία δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια με την Επιτροπή των Προπολογισμών. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τους ε, οργανισμούς, όχι καθέναν βέβαια ξεχωριστά, αλλά ε, να σας πω εν γέννη τι είναι αυτό το που προσθέτουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να σας ενημερώσω για τις δράσεις που έχουμε αναλάβει από πέρυσι σε αυτό το ίδιο πλαίσιο και τις προκλήσεις ε, τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε με βάση το ε, προτινόμενο προϋπολογισμό καθώς και τις βλέψεις μας για το μέλλον. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι πολύ σημαντικοί συνιστόσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δημιουργούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα για να εκπονήσουν νομικά, τεχνικά ή επιστημονικά καθήκοντα. Εμείς, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, ε, θα δίνουμε συμβουλές ώστε να σχηματιστούν ε, νήμερα οι πολιτικές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Διεξάγουμε αξιολογήσεις κινδύνου αλλά και εποπτικές λειτουργίες καθώς και λειτουργίες πιστοποίησης. Εντοπίζουμε, αξιολογούμε και επικοινωνούμε όσον αφορά τις υφιστάμενες αλλά και τις αναδυόμενες απειλές πολλές. Εξυπηρετούμε τους πολίτες προωθώντας την ε, ε, διάδοση των πληροφοριών ε, όσον αφορά τα πορίσματά μας σε πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. οργανισμοί όπως το Food and Drug Administration στη ΣΥΠΑ έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν ειδικευμένες συμβουλές στις εθνικές τους κυβερνήσεις. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν παρομοίω για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών πιο αποτελεσματικά και για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες που εντοπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη. Εργαζόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα ε, θεμάτων που αγγίζουν τις ζωές ε, καθενός ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, ε, επί της γης, στις θάλασσες αλλά και ακόμα στον αέρα. Καλύπτουμε τα φάρμακα, τα χημικά, την παιδεία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια και φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι βέβαια πλήρης, αλλά απλά σας δίνει μια γεύση για τις πολλές ειδικευμένε ε, ασχολίες μας οι οργανισμοί δεν είναι μόνο ουσιαστικοί για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων, αλλά διευκολύνουν επίσης ε, να γίνουν οικονομίες κλίμακας σε πολλούς τομείς, καθώς οι οργανισμοί μειώνουν το συνολικό κόστος για τους φορολογούμενους. Για να το πω πιο απλά, συχνά είναι φθηνότερο να κάνει κανείς κάτι ε, μια φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά να το κάνει 28 φορές σε εθνικό επίπεδο. Οι οργανισμοί καταναλώνουν ε, τη σήμερα συνολικά 0,6% του συνόλου του ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Πριν από αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να έχετε λάβει, όπως είπατε, Πρόεδρε, από πλευρά μας ένα έγγραφο που περιλαμβάνει σύντομα ε, τις βασικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί αν περάσει η πρόταση προϋπολογισμού 2015 ως έχει. Να σας δώσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Η διαδικασία προϋπολογισμού για το 2015 λαμβάνει χώρα όταν οι υπουργοί των, μάλλον πολλά κράτη των κρατώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ε, πολλές δυσχέρειες και δημοσιονομικούς περιορισμούς. Επειδή οι οργανισμοί δεν είναι τοποθετημένοι στα κράτη-μέλη κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, κατανοούν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πριν λοιπόν να μπω σε πιο λεπτομερείς συζητήσεις για τις προτάσεις ε, ε, της Κομισιόν όσον αφορά την ε, χώρεση πόρων των οργανισμών, θα ήθελα να τονίσω πως οι οργανισμοί είναι απόλυτα προσιλωμένοι στο να προσφέρουν το δικό τους μερίδιο ανάλογα με τα μέτρα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η δύσκολη, η δυσχερή σε αυτή η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα. Τούτου λεχθέντος, οι οργανισμοί ενεργά εξετάζουν τις δυνατότητες επεκτηνόμενων περιοχών συνεργασία αύξησης της διαφάνειας και τέλος αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητα. Αυτό το κάνουμε εισάγοντα σύγχρονε τεχνολογίε στη δημόσια διοίκηση, καθώ και αποτελεσματικά εργαλεία όπω ε, ε, ο προπολογισμό με βάση τι δραστηριότητε, διαχείριση με βάση τι δραστηριότητε και ε, κοστολόγηση με βάση τι δραστηριότητε. Αυτά είτε έχουν ήδη εφαρμοστεί είτε εφαρμόζονται, είναι στην πορεία της εφαρμογής, έτσι ώστε οι οργανισμοί να εξετάσουν όλες τις πιθανότητες για εξορθολογισμό και εξοικονομήσεις. Οι οργανισμοί σέβονται την απόφαση που έλαβαν από κοινού Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν στη κοινή δήλωση και κοινή προσέγγιση από το 2012 καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες ε, της ε, Κομισιόν μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε όσον αφορά την εφαρμογή του δικού χάρτη για την ε, συνέχεια πρέπει να δοθεί στην κοινή προσέγγιση. Οι δράσεις κλειδιά του δικού χάρτη έχουν στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οργανισμών και τη λογοδοσία τους. Ο δικός χάρτης έχει στόχο την εισαγωγή μεγαλύτερη συνοχή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί και οι περισσότερες δράσεις έχουν ήδη εφαρμογιστεί και θα, οριστικό, θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του έτους, προσφέροντας έτσι περισσότερη ακόμα αποτελεσματικότητα. Παρά όμως όλες αυτές τις ενέργειες τις οποίες έχουν προβεί οι οργανισμοί, δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τις περικοπές που επιβάλλει η Κομισιόν σε μας, όπως αυτές, ιδιαίτερα μάλλον για τους οργανισμούς που έχουν πια φτάσει την ταχύτητα κρουαζιέρας τους, που έχουν δηλαδή μπει σε ένα κανονικό ρυθμό λειτουργίας. Η συμφωνία προβλέπει ως στόχο την σταδιακή μείωση του προσωπικού σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και στους οργανισμούς και σώματα, κατά 5% σε διάστημα 5 ετών. Για το σημείο αυτό θα ήθελα σαφώς να δηλώσω πως ε, οι οργανισμοί όχι μόνο δέχτηκαν αυτή τη μείωση, αλλά οι περισσότεροι με μεγάλη όμως δυσκολία το έχουν εφαρμόσει μέσα στην πολιτική, στα πολιτικά τους προγράμματα για το, την επόμενη πενταετία όσον αφορά το προσωπικό. Όμως αυτά τα οποία προβλέπει η Κομισιόν ε, επιβάλλουν περαιτέρω περικοπή πέρα από το 5% και για τους ε, οργανισμούς που λειτουργούν με κανονικό ρυθμό επιβάλλουν ε, ακόμα περισσότερη μείωση για τη δημιουργία αυτού του πουλ αναδίπλωσης. Το είδαμε αυτό και στην ανακοίνωση του Ιμπερσινή, την ανακοίνωση που το ίδιο το Κοινοβούλιο την απέρριψε. Όπως και το Κοινοβούλιο, οι οργανισμοί διαφωνούν κάθετα με αυτή την πρόταση. Η προσέγγιση της ε, DG Budget είναι να ε, θεωρήσει τους πόρους όλων των οργανισμών ως ένα κονδύλι. Δηλαδή, όταν ένας οργανισμός παίρνει επιπλέον πόρους για να εκπληρώσει την νομική της εντολή ή όταν δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός, άλλοι οργανισμοί ταυτό, ε, αυτομάτως βλέπουν τους δικούς τους πόρους να περικόπτονται. Η γραμμική αυτή προσέγγιση στο περικοπή κατά 5% έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις. Ε, οι περισσότεροι, πιο παλιοί οργανισμοί λοιπόν χρειάστηκε να εφαρμόσουν όχι 5% μείωση προσωπικού αλλά 10% μείωση προσωπικού. Αυτό δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλο ίδρυμα ή σώμα. 10% δεν είναι το 5% που συμφώνησαν ε, ε, μέσω της διοργανικής συμφωνίας. Αυτό προτείνεται χωρίς άλλη αποζημίωση, ούτε από τη μορφή μείωσης ε, των επιβαλλόμενων νομικών υποχρεώσεων για την εκπόνηση ορισμένων καθηκόντων, ούτε μέσω αύξηση του προπολογισμού που θα επέτρεπε ένα επίπεδο outsourcing για τα ε, καθήκοντα τα οποία δεν είναι τα πιο ουσιαστικά. Πρόκειται για άνηση μεταχείριση. Οργανισμοί με ε, ιδρύματα από τη μια πλευρά και παλιοί οργανισμοί απέναντι σε νέους οργανισμούς με νέα καθήκοντα να σας ε, δώσω ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν με συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ποιο είναι το σχήμα που ακολουθείτε. Δηλαδή, το παράδειγμα του, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Αεροπλοεία. Η Κομισιόν έχει καθορίσει αυτόν τον οργανισμό ως οργανισμό με νέα καθήκοντα. Προβλέπονται 693 θέσεις για το 2015. Από αυτές, 463 χρηματοδοτούνται από τα τέλη και τις χρεώσεις. Οι υπόλοιπε θέσεις πληρώνονται από τον προπολογισμό της Ένωσης. Λόγω νέων καθηκόντων, αυτός ο οργανισμός ζήτησε αύξηση 8 από τις χρηματοδοτούμενες, τις επιδοτούμενες θέσεις. Η Κομισιόν συμφωνεί, αλλά ταυτόχρονα προτείνει μείωση 14 θέσεων που χρηματοδοτούνται από, χρέη και τε, από χρεώσεις και τέλη. 8 νέες θέσεις προς 14 λιγότερες περικοπές. Οι 14 αυτές θέσεις είναι μέσα στο όριο προσλήψεων. Δεν είναι στόχος. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, αυτό εξαρτάται από το φόρτο εργασίας και από τη ζήτηση. Με λίγα λόγια δηλαδή, οι περικοπέ δεν πρέπει τυφλά να εφαρμόζονται χωρί να λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσει, όπω στην περίπτωση του οργανισμού ε, αεροπλοεία που χρειάζεται κάποια ευελιξία ώστε να μπορεί χρονικά να ανταποκρίνεται στα αιτήματα επαληθεύσεων που προέρχονται από τη βιομηχανία αεροπλοεία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή, θα ήθελα να σα πω ότι Ήδη χρησιμοποιούμε τις ε, δυνατότητές μας μέχρι ε, τα... έχουμε φτάσει στα όρια μας. Οι προκάτοχοί μας ε, στους οργανισμούς είχαν προειδοποιήσει την Κομισιόν για όλα αυτά και αυτό γίνεται πλέον πραγματικότητα. Οι οργανισμοί πρέπει πλέον να, να συμπτύξουν τις δραστηριότητές τους διότι δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους για να τις φέρουν εις πέρας. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι αυτό ίσχυε πριν από δύο χρόνια ήδη, όπου μόνο ένας οργανισμός δεν μπορούσε να αναλάβει ένα καθήκον και το οποίο προβλεπόταν νομικά, ενώ τώρα αυτό έχει γίνει πια κοινό τόπος ε, για όλους τους οργανισμούς σχεδόν. Ωστόσο, όλα ένα περισσότερα ζητάει ε, κοινοτική νομοθεσία από τους οργανισμούς να κάνουν. Πολλά από τα νέα καθήκοντα, επιχειρησιακά αλλά και διοικητικά, ξεπερνούν τις νομικές πράξεις. Μάλιστα τα νέα καθήκοντα πολύ συχνά είναι πιο σημαντικά από την εξέλιξη των υφισταμένων καθηκόντων. Οι οργανισμοί συχνά πέφτουν θύματα της επιτυχίας τους, πράγμα που σημαίνει ότι όσο καλύτερη είναι η αποτελεσματικότητά τους, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση από αυτές. Ωστόσο, αυτά, σε αυτά πρέπει να ανταποκριθούμε με λιγότερους πόρους. Συγκεκριμένα παραδείγματα φυσικά θα βρείτε στο σημείωμα που σας έχουμε ήδη δώσει. Όμω στην ουσία αυτό δεν μπορεί επαόριστο να συνεχίζεται και οι οργανισμοί όλα ένα και συχνότερα αντιμετωπίζουν το δίλημα πώς θα μπορέσουν σωστά να ανταποκριθούν στην εντολή τους με τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι σωστό οι διευθυντές των οργανισμών και τα διοικητικά συμβούλια να αναγκάζονται να αποφασίζουν ποιο κομμάτι της εντολής τους θα ε, ε, ε, υλοποιήσουν. Οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να παραβλέπουν καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από εσά, τους νομοθέτες, του ιδρυτικού μας κανονισμού ή του καταστατικού μας ή άλλων νομοθεσιών που επηρεάζουν τις δραστηριότητε μας. Ξέρω πως πολλοί διοικητές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντέ είναι, αισθάνονται πολύ άσχημα με αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευθούν μέσω της σωστής αξιολόγησης των αναγκών κάθε οργανισμού, ανά περίπτωση, ε, σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντι, της αντίστοιχης ε, πολιτικής, του αντίστοιχου τομέα πολιτικής. πρέπει να ληφθεί υπόψη η εντολή του οργανισμού και ο συσχετισμός των καθηκόντων ε, του προσωπικού του κάθε οργανισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν κάθε φορά. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε ως σημείο κίνησης για να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις περί Γνωρίζουμε ότι αν εξεταστεί ο κάθε περίπτωση ξεχωριστά, και αν ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες για καθέναν οργανισμό μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια από τους οργανισμούς αλλά και από τις αρχές ε, τις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, λογικές αλλά και βιώσιμες εξοικονομήσεις. Η βάση για αυτή την προσέγγιση υπάρχει ήδη όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ειδικευμένες του επιτροπές αντέλαξαν ε, πληροφορίε με του οργανισμού για την εντολή του, εξέτασαν τα προγράμματα εργασία του και ε, πρόσφεραν τι ειδικευμένε του νομοδοτήσει στην Επιτροπή Προπολογισμού κατά τη διάρκεια τη δημοσιονομική διαδικασία. Πιστεύω πω αυτή η αναπερίπτωση εξέταση μπορούσε να ενισχυθεί μέσω ετούτη εδώ τη επιτροπή, ώστε να προσαρμοστεί ο προπολογισμό, αλλά και τα προγράμματα ε, ε, ε, πάνω σε εξολογημένε ανάγκε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή που αναγνωρίζει τη σοβαρότητα αυτών των θεμάτων και που εξακολουθεί σταθερά να στηρίζει τις, ε, τους οργανισμούς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και όλο ιδιαίτερο να ευχαριστήσω για τις ξεκάθαρες δηλώσεις τις οποίες προέβη το Ευρωκοινοβούλιο και τούτη η Επιτροπή στις γενικές του κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία και την κατάρτιση του προπολογισμού 2015. Υπογραμμίζεται εκεί την ανάγκη να αξιολογηθούν όλοι οι οργανισμοί αναπερίπτωση όσον αφορά τον προπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους τους. Τώρα, για το μέλλον θα ήθελα να ολοκληρώσω μιλώντας σας για το νέο διαθεσμικό, θεσμική ομάδα εργασίας. Εμείς ε, καλωσορίζουμε τη δημιουργία αυτής της ομάδας εργασίας που θα εξετάσει τους πόρους των ε, αποκεντρωμένων οργανισμών με στόχο να βρει ε, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τους οργανισμούς με βάση αντικειμενικά κριτήρια και αξιολογικά κριτήρια. Χαίρομαι που βλέπω το ενδιαφέρον του νομοθέτη για το μέλλον των οργανισμών. Πιστεύω στεναρά και οι συνάδελφοι εδώ νομίζω θα συμφωνούν επίσης ότι θα πρέπει αυτοί οι οργανισμοί να εξεταστούν μεμονωμένα αλλά και ως ένας μηχανισμός στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης επί τη βάση της εμπειρογνωμοσύνης από την καθημερινή μας εργασία μέσω των 30 και πάνω οργανισμών που υπάρχουν σε ολόκληρη Ευρώπη. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα και να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις. Έχουμε πολλές ιδέες στο δίκτυο και διαφθορτικές ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία των οργανισμών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς αυτό, χωρίς μάλλον να, να, να παραβλέψουμε τις, ε, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, γιατί δεχόμαστε την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντική η εργασία τη ομάδα εργασία για τους οργανισμούς γιατί επηρεαζόμαστε άμεσα από τα απορίσματα της ε, ομάδας εργασία. Οι οργανισμοί λοιπόν γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν και είμαι πεπισμένος ότι οι οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν προς όφελος όλων των μερών. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη ε, επαφή, ε, αλληλεπίδραση. Είμαστε στη διαθεσή σας ε, ως πρόεδρος του δικτύου, αλλά και όλοι οι οργανισμοί είναι στη διαθεσή σας για να στηρίξουν την ομάδα εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε, Αντιπρόεδροι, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτές που ακούσατε την εισήγησή μου και με χαρά προσβλέπω στη συνεχιζόμενη συνεργασία με την Επιτροπή σας ε, στη διάρκεια των δύσκολων χρόνων που μας περιμένουν. Και φυσικά προσβλέπω στις ερωτήσεις, στα σχόλιά σας και οι συνάδελφοί μου από τους οργανισμούς είναι επίσης ε, στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. έχει να προσθέσει κάτι μήπως ο Μαρσέλ από τον Οργανισμό για την Κατάρτιση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι Μάρτιν τα είπε πραγματικά πολύ ξεκάθαρα και ίσως είναι προτιμότερο να περιμένω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Εννοείται ότι ο συντονισμός των οργανισμών, το συντονιστικό όργανο των οργανισμών θα σας προσφέρει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε, είτε δεδομένα βάσης, είτε και οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των προϋπολογισμών μας. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κύριε Καρούν, έχετε προσέλθει συνοδευόμενος από πολυάριθμους συναδέλφους σας, οι οποίοι αν θέλουν να συμπληρώσουν τα λόγια σας, ευχαριστώ να τους ακούσουμε. Αν δεν υπάρχει επιθυμία λήψεως ε, λόγου από πλευρά των συναδέλφων σας, ίσως μπορούν να απαντήσουν αργότερα στις ε, παρατηρήσεις που θα κάνουν οι συναδελφοί μου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Monsieur Λέγομαι Ζδεχόσκι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρέμβασή σας. Έχω βεβαίως ε, μεγάλο σεβασμό για το έργο των οργανισμών. Θα ήθελα όμως να εκφράσω και την εντύπωση που έχω ως νέος Ευρωβουλευτής ότι όταν μιλούμε για τέτοια θέματα θα πρέπει να είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι. Είπατε ότι προδιετίας Ένας μόνο οργανισμός δεν μπόρεσε λόγω περικοπών να εκπληρώσει την εντολή της. Δηλαδή ότι τώρα μετά από μια διετία είναι πάρα πολλοί οι οργανισμοί που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις εντολές τους. Όταν κάποιος τοποθετείται τόσο αόριστα, εμένα μου προκαλεί ένα περίεργο συνέστημα. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς πόσοι οργανισμοί δεν μπορούν να εκπληρώσουν πλήρως την εντολή τους και γιατί όχι. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω στις απαντήσεις σας να προχωρήσετε σε λεπτομέρειες. Δεν μπορώ αλλιώς να έχω εικόνα για το πόσα από τα όργανά σας έχουν προβλήματα και για ποια πόσα πρόκειται. Αν συμφωνείτε, λέει ο Πρόεδρος, θα ακούσουμε έναν αριθμό παρεμβάσεων και μετά θα απαντήσετε σε όλες μαζί. Ας ακούσουμε μια πρώτη σειρά πέντε παρεμβενόντων. Κύριε Γκάιερ, εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς τους οργανισμούς και άλλη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα, οργανισμοί. Σωστά είπατε ότι το τμήμα εκείνο του προϋπολογισμού που σας αφιερώνεται είναι σχετικά περιορισμένο σε σχέση με τις διαστάσεις των ποσών που έχουμε συνήθως όταν παρακολουθώ την δημόσια συζήτηση για τους οργανισμούς και στην πατρίδα μου, τη Γερμανία, μπορεί κανείς τότε να αποκομίσει την εντύπωση ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέσει σαν τα κοράκια πάνω στον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται με το τίποτα άλλο με το να αυξάνει τον αριθμό τους. Μιλάμε όπως είπατε και εσείς για 0,6% του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ίσως αυτό να τρομάξει κάποιους δημοσιογράφους ως ποσοστό και είπατε και σωστά εσείς επίσης ότι ορισμένοι από τους οργανισμούς σας λόγω της μεταχείρισης που τους επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν φτάσει στο χείλος της μη δυνατότητας λειτουργίας. Εμείς θα θέλαμε πάντως το σημερινό απόγευμα να εγκύψουμε στην υπόθεση αυτή. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό θα κάνουμε. Ωστόσο, η ερώτηση που διατυπώνω έχει ως εξής. Κατά πόσο συζητείτε τα προβλήματα αυτά με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί αυτές είναι που θα μας υποβάλουν μετά γνωμοδοτήσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, σε εμά εδώ την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρόσκληση λοιπόν δική μου είναι να πάτε στις ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές που γνωρίζουν και εκτιμούν καλύτερα το έργο σας, να ζητήσετε εκεί την υποστήριξη των μελών τους και μέσω των γνωμοδοτήσεων που υποβάλλουν αυτές οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης που θα εξοπλίσουν νομοδοτήσεις αυτές και με τα σχόλια που θα υποβάλλετε, νομίζω ότι θα αποδώσουν πολύ περισσότερο από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε να, να συζητήσουμε μεταξύ σας. Βεβαίως δεν θέλω να πάυσει αυτή η επαφή που έχουμε μαζί σας. Θέλω να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των οργανισμών, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας αλλά σας υποδεικνύω πού θα πρέπει καταρχήν να βρείτε συμμάχους μέσα στο ε, σώμα, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, Κομισιόν, μπορούν οι οργανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Για πέντε χρόνια ήμουν συντονιστής της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Του προϋπολογισμού. Είναι δηλαδή η Επιτροπή εκείνη η οποία συζητεί την ετήσια απαλλαγή του προπολογισμού των οργανισμών. Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, καμιά φορά ζήσαμε και πολύ έντονε συζητήσει και αντιπαραθέσει γύρω από το ερώτημα εάν στους επιμέρους οργανισμούς γίνεται σωστή χρήση των πόρων της Ένωσης. έγινε και η πρόταση και υπήρξε συμφωνία να υπαχθούν οι οργανισμοί σε οικονομικό έλεγχο εξωτερικό. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει τον έλεγχο αυτόν. Έχω τώρα την Common Approach του 2012, την οποία εγώ ερμηνεύω έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει θα υποστηρίξει τους οργανισμούς για να ψάξουν να βρουν αυτό τον εξωτερικό οικονομικό ελεκτή Ότι δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να το πράξει αυτό. Αυτό είναι για μένα σαφέ. Διότι τότε θα έπρεπε να παραιτηθεί από την ανεξαρτησία του. Όμω το συνέδριο μπορεί να υποστηρίξει τους οργανισμούς να αναζητήσουν και να εξεύρουν οικονομικό ελεγκτή. Βλέπω τώρα, διαβάζω τώρα ότι τον Ιούνιο Φέτο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να μεταφέρουν το καθήκον αυτό στους οργανισμούς. Ωραία, καλά κάνει τώρα η Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο γιατί έτσι ξεμπερδεύουν το πρόβλημα και με τη χρηματοδότησή του. Αλλά δεν βελτιώνει όμω ούτε διευκολύνει την θέση των οργανισμών. Διότι ο πυρήνα τη εντολής των οργανισμών δεν είναι να βρουν τον ε, εξωτερικό οικονομικό ελεγκτή. Το έργο του είναι να συμβουλεύουν τον νομοθέτη. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιοι λόγοι την παρακίνησαν να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο για την επίλυση του προβλήματος της εξέβρεσης του auditor. Με όλα όσα σημαίνουν προκηρύξεις, ε, προσκλήσεις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και Όλα αυτά λοιπόν να τα μετακυλήσουν στους οργανισμούς. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση, κάπως γενική. Διαβάζοντας το έγγραφο θέσεων των οργανισμών, βλέπω ότι επιμένουν διαρκώς επί της ανάγκης όσον αφορά την κατανομή πόρων να εργαστούμε σε μια περιπτωσιολογική προσέγγιση, σε μια περιπτωσιολογική βάση, case by case. ώστε να καταλήξουμε στην δυνατότητα ενδεχομένω 5% περικοπών. Η ερώτησή μου είναι εξή τώρα. Πρώτα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η γνώμη της Κομισιόν για την πρόταση αυτή που κάνουν οι οργανισμοί. Και ιδίω την σύσταση που κάνουν στο έγγραφο αυτό στη σελίδα 8 όπου λένε ότι θέλουν να δουλέψουν πάνω σε μια βάση case by case και κάνουν εκεί τρεις συστάσεις. Αυτές οι συστάσεις είναι συμβατές, άραγε με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε λοιπόν με αυτή την case by case ο κ. Ντεπρέ γυρνά μακριά από το μικρόφωνο, στρέφεται προς τα πίσω και δεν τον ακούμε. Τώρα ακούγεται καλύτερα. Πώ μπορούν να επιτύχουν λοιπόν του αντικειμενικού σκοπού, Αυτό θα ήθελα να μάθω. Ο κύριος Μάνκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Το ελεγκτικό συνέδριο προ 12-13 ετών είχε κάνει μια ανεξάρτητη audit για τον εαυτό του. Ήταν ο πρώτος τότε ε, οικονομικός ε, έλεγχος και έκτοτε έχουν επιτύχει κάθε έτος να μειώνουν το κόστος. Αποδοτικότερη λοιπόν η προσπάθεια κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν. Εάν προσφέρουμε τη δυνατότητα εξωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς, θα υπάρξει δυνατότητα βελτίωσης. Παντού χωρί βελτίωση. Άλλοι θα έχουν δυνατότητα βελτίωση 20%, άλλοι θα έχουν δυνατότητα βελτίωση 2%. Εγώ έχω εμπειρία με τη διαχείριση οργανισμών ή οργανώσεων και πάντοτε είχαμε βρει τη δυνατότητα να βελτιωθούμε. Κάντε λοιπόν ό,τι μπορείτε καλύτερο. Αν όμως δεν έχουμε στα χέρια μας επιχειρήματα, δεν μπορούμε να δείξουμε και τρόπους βελτίωσης. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος και αυτός θα σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι πρέπει να ποσοτικοποιηθούν όλες οι απαιτήσει σας και να υποβληθούν από πλευρά σας δηλαδή των οργανισμών στις ε, αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εκεί τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα σας δώσουν συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν στις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες είμαι βέβαιος θα σας υποστηρίξουν. Και εφόσον είναι δικαιολογημένα τα αιτήματά σας, θα σταθούν δίπλα σας. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Αλλιώς θα είναι υπερβολικά υποκειμενική οποιαδήποτε τοποθέτηση κάνουμε τώρα. Ο κύριος ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος των αποκεντρωμένων οργανισμών σχολίασε τα περί τρέχοντος προπολογισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι δεδομένου του έργου τους είναι σαφές που το έθεσε έτσι όπως το έθεσε. Εγώ δεν μπορώ βέβαια να είμαι ουδέτερος, αλλά θέλω να τον ρωτήσω το εξή. Οι περικοπές που προβλέπονται στον προπολογισμό και στο προσωπικό των οργανισμών έχουν να κάνουν με τεχνικά δεδομένα, δηλαδή περίσευαν πόροι από τους οργανισμούς ή οφείλεται αυτό σε περισσότερο ιδεολογικού χαρακτήρα λόγους. Δεύτερον, ακόμα και αν ισχύει ότι υπήρχε πλεόνασμα πόρων στους οργανισμούς, που θα μπορούσε ίσως, θα ήθελα να το μάθω. Και είναι λογικό στην κατάσταση αυτή κοινωνικής κρίσης που βρισκόμαστε να έχουμε αύξηση στους οργανισμούς για την ασφάλεια και την αστυνομία και περικοπές στην τεχνολογική έρευνα, το περιβάλλον, μεταφορές, συνθήκες εργασίας είναι φυσικό αυτό, σας φαίνεται φυσιολογικό αυτό στις εποχές που ζούμε. Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές ότι θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ασφάλεια στην Ευρώπη από ό,τι τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάποιος έκτος έχει ζητήσει το λόγο, θα τον προσθέσουμε. Παρακαλώ, ε, κύριε Σκόλμελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα για τις πραγματικά πολύ λεπτομερείς τοποθετήσεις. Μέχρι τώρα εργαζόμουν στο ελεγκτικό συνέδριο της Βάδης Βιτεμβέργης. Εκεί έχουμε κάνει κατ' επανάληψη έρευνες για την χρησιμότητα, λειτουργία ε, δημοσίων υπηρεσιών και αρχών. Κάθε μια από αυτές βεβαίως μπορεί να εξηγήσει και να ορίσει γιατί είναι απαραίτητο το έργο της. Εκεί μάλιστα οι όλοι οι αξιωματούχοι είναι ε, εξαιρετικά επιμελείς και αν τους αφήσετε μόνους τους κάθε χρόνο θα σας υποβάλουν όλο και περισσότερα αιτήματα. Εδώ για τους οργανισμούς προβλέπουμε 0,6% για το προσωπικό τους, της 100 του προϋπολισμού. Μιλούμε όμως και για 6.000 θέσεις οργανογράμματος, οργανικές θέσεις δηλαδή, μοιρασμένες σε 32 οργανισμούς. Θα έπρεπε εδώ πρώτα να γίνει μια ανάλυση των καθηκόντων. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε 32 οργανισμούς, 32 οργανικές ενότητες, Όντως το έργο τους προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία. Όντως είναι απαραίτητες υπερεθνικά. Γίνεται δηλαδή κάποια εξοικονόμηση στο εθνικό επίπεδο λόγω της ύπαρξής τους. Και αυτές οι οργανικές ενότητες είναι έτσι δομημένες ώστε όντως το έργο τους να περιορίζεται στο ουσιώδες. Εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Είτε έχω ένα συγκεκριμένο κονδύλι και θέλω να το χρησιμοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο, είτε έχω μια συγκεκριμένη χρήση και λέω θέλω να την επιτύχω, να λειτουργήσει δηλαδή αυτό που θέλω, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η δεύτερη παραλέγη είναι αυτή που πρέπει να ισχύει σήμερα, δηλαδή πρέπει με το δυνατόν λιγότερα κονδύλια να μπορούμε να επιτύχουμε ένα δεδομένο όφελος. Ο Πρόεδρος, δεν ε, έχω άλλες αιτήσει λήψεως του λόγου. Εγώ είμαι βέβαια καινούριο εδώ στην Ευρωβουλή και βέβαια στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ένα θέμα. 32 οργανισμοί, αλλά στον κατάλογο που μας έχετε κοινοποιήσει, που λέει ε, έγγραφο θέσεων του δικτύου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, βλέπω 41 δομές. 32-41 υπάρχει μια διαφορά. Έχω σημειώσει ότι ζητείτε να γίνει μια ανάλυση κατά περίπτωση. Δεν μπορούν άραγε να διακριθούν οι οργανισμοί ανα είδος, δηλαδή υπάρχουν ρυθμιστικοί οργανισμοί, για παράδειγμα χρηματοπιστωτικές αγορές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ε, πρόνοιας, για την ε, ε, διάλυση των τραπεζών ενδεχομένω. Επομένως, οι οργανισμοί αυτοί είναι ανεξάρτητες αρχές. Από την άλλη μεριά, στην βάση ενδεχομένως όπου το Κοινοβούλιο θα καθορίσει το έργο τους. Υπάρχει λοιπόν ένα, ένας χώρος ιδίων πόρων, δηλαδή για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για έναν αριθμό οργανισμών. Και ίσως μπορεί να γίνει η διάκριση αυτών των οργανισμών από άλλους που έχουν περισσότερο λειτουργία παροχή συμβουλών προς το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κολμέλ σε ένα σημείο. Ίσως υπάρχει μάλιστα επικάλυψη στο έργο ενός ευρωπαϊκού οργανισμού και, και εθνικών αρχών. Ίσως ορισμένες χώρες μέλη όντως με την ύπαρξη των οργανισμών να κάνουν κάποιες εξοικονομήσεις. Ίσως να μην χρειάζονται τότε κάποιοι εθνικοί οργανισμοί εάν το έργο που γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υποκαταστήσει κάποιο μέρος του έργου που γίνεται στο εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό το συγκεκριμένο. Και επίσης, συνολικότερα, αν χρειάζεται να γίνει οικονομική έλεγχη ανά οργανισμό, πως χρειάζεται και ένας έλεγχος για το σύνολο των οργανισμών, για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επικαλύψεων, ιδίω να δημιουργηθούν κάποιοι πυρήνες οργανισμών, κάποια κλάστερ. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που είχα εγώ με τη σειρά μου. Θα δώσουμε το λόγο τώρα με τη σειρά στον κύριο Κερούν πρώτα, αν συμφωνεί, και μετά στον Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Προϋπολογισμών της Κομισιόν, κύριο Κεσάν. Βεβαίως στην, στις απαντήσεις σας μπορείτε να έχετε και την συμβολή των συναδέλφων σας που είναι μέλη της Τρόικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα τόσο πλούσια σχόλια, αλλά και τις ερωτήσεις που υποβάλλατε στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Όλα αυτά είναι πολύ υποσχόμενα για τον συνεχιζόμενο διάλογο ανάμεσα στους οργανισμούς και την Επιτροπή σας προσβλέπουμε να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο μέσα στους επόμενους μήνες και χρόνια. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με εσά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που ρωτήσατε για το 42 και το 31. Κοιτάξτε, στο δίκτυο των οργανισμών έχουμε και τις ε, κοινέ συμπράξεις. Η καθαρή εθέρες, για παράδειγμα, που είναι το πιο πρόσφατο μέλος στο δίκτυό μας για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή, επιπλέον ομάδας που υπάρχει με δομή σε των οργανισμών. Γι' αυτό και τους έχουμε συμπεριλάβει και αυτούς στο δίκτυό μας όσον αφορά τις άτυπες ανταλλαγές απόψεων που έχουμε. Τα άλλα δύο θέματα που τέθηκαν τώρα. Κατά πόσο είναι εφικτό να βάλουμε μαζί τους οργανισμούς, να τους ομαδοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Κοιτάξτε, θα γίνει ο διάλογος αυτό στους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν στην τρέχουσα κατάσταση για τους οργανισμούς. Είπατε κι εσείς αν υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε μαζί κάποιους οργανισμούς ή αν θα μπορούσαν να προσελκύσουν εξωτερική χρηματοδότηση κάποιοι οργανισμοί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλά τέτοια ζητήματα που τίθεται, αλλά θα τα εξετάσουμε περίπτωση κατά περίπτωση για να εντοπίσουμε νέους τρόπους χρηματοδότησης. Υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στους οργανισμούς με πολλούς και διάφορους τρόπους. μία, ένας οργανισμός μπορεί να έχει αναπτύξει πολύ πιο προχωρισμένες μεθόδους διαχείρισης από ότι κάποιος άλλος οργανισμός είτε για την πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τους διαγωνισμούς δηλαδή, είτε για οτιδήποτε άλλο. Οπότε υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους για θέματα προσωπικού, για παράδειγμα, αλλά και άλλα. Αλλά και αυτό μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος στα ονόματα. Ο κύριος Σακόφσκι ήταν νομίζω. Για την ιδιαιτερότητα. Στο σημείωμα που σας δώσαμε θα δείτε στο παράρτημα διάφορα παραδείγματα οργανισμών. Γίνεται συντονισμός, κάνουμε έρευνες Άμα θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ αναφέρονται μόνο κάποια παραδείγματα οργανισμών. Αλλά ίσως οι συνάδελφοι που είναι εδώ να μπορούν να πούνε περισσότερα. Είτε για τον Οργανισμό για τα Ναρκωτικά στη Λισαβόνη είναι εδώ ο συνάδελφος. Άμα θέλετε θα μπορούσε να σας πει μετά ποιε είναι οι επιπτώσεις. Και εγώ από το δικό μας τον οργανισμό μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τα καθήκοντά μας και για τους εννέα τομείς που μας απασχολούν, δεδομένου ότι δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση. Ευχαρίστω πάντως να επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Για τον κύριο Γκάιερ. λέτε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την προστιθέμενη αξία. Πού είναι αυτή η προστιθέμενη αξία. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό οι οργανισμοί ακριβώς για να δούμε αν οργανισμό αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το προφίλ των οργανισμών που αυτό θέλετε, γιατί ρωτάτε τι κάνουν αυτοί οι οργανισμοί, πώς μπορούν να γίνουν πιο ορατοί, πώς μπορεί να προβληθεί η δουλειά τους περισσότερο προς τα έξω. Πώς θα γίνει ο κόσμος να ξέρει τι προσφέρουν. Επίσης και το άκουσα αυτό στην ερώτησή σας, λέτε πώς εμείς στο εσωτερικό μας μπορούμε να συζητήσουμε για να ενισχύσουμε και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Είναι και αυτό κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε και περιλαμβάνεται στο διάλογο που έχουμε μαζί σας. Και θα ήθελα να ακούσουμε από εσά περισσότερα να έχουμε τέτοιες ε, συναντήσεις πιο συχνά για να ακούμε και τις δικές σας τις ιδέες, όπως επίσης να ξέρουμε και τι περιμένουν οι χώρες μέλη από τους οργανισμούς μας. Στον κύριο Ντεπρέ τώρα να απαντήσω. λέτε πώς θα, γίνει, πώς θα γίνουν οι περικοπές. Είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί αυτό. Και γι' αυτό και θέλουμε να εξετάσουμε αναπερίπτωση τον κάθε οργανισμό, την κάθε ομάδα, τον κάθε τομέα, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην οροφή, στόχο που είναι 5% ή ό,τι και αν είναι και πώς μπορεί να συνεισφέρει αυτό. Οι οργανισμοί δεν αντιτίθεται, δεν αντιστέκονται. Απλώς θέλουμε να δούμε πώς μπορεί καλύτερα να γίνει αυτό από εμά, από άλλα όργανα. Στο διάλογο αυτό Πάντως με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θέλουμε να έχουμε και διάλογο για τις προτεραιότητες. Όπως είπα και στην αρχή, και οι διευθυντές και τα διευθυντικά συμβούλια το βρίσκουν κάπως περίεργο γιατί έχουμε νομική υποχρέωση να κάνουμε κάτι και πώς είναι δυνατόν αυτό να το παρακάμψουμε. Και θέλουμε να το συζητάμε αυτό με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στον κύριο Μάνκα, να απαντήσω τώρα για τον ανεξάρτητο έλεγχο και πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί πάλι. Γίνεται πολύς έλεγχος στους οργανισμούς και υπάρχει διαφάνεια. Αν μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα αυτό, ευχαρίστως να μας συμβουλεύσετε. Να ξέρετε πάντως ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι στη δουλειά μας και όσον αφορά τη διαχείριση, διακόπτει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι ο κύριος Ντεπρέ θέλει να αντιδράσει σε αυτό που λέτε. Του επιτρέπετε να σας διακόψει για να σας ρωτήσει κάτι. Ναι. Λοιπόν, στην ε, κατά περίπτωση προσέγγιση, έτσι, και βασίζομαι εδώ στο έγγραφο το οποίο μας ε, δώσατε. Καταλαβαίνω πολύ καλά το κατά περίπτωση. Θέλετε κατά περίπτωση λοιπόν να σεβαστείτε το αυτόνομο καθεστώς ε, των οργανισμών, μια που με διαφορετική πράξη ιδρύθηκε ο καθένας από αυτούς. Πολύ ωραία. Έχουν λοιπόν ο κάθε οργανισμός μια ιδιαιτερότητα. Και είναι και κάποιες που δημιουργήθηκαν χωρίς καν να έχουμε συμφωνήσει εμείς. Αλλά λέτε ότι με την καταπερίπτωση προσέγγιση θα καταλήξετε για τον κάθε οργανισμό στο ίδιο αποτέλεσμα που θέλει η Επιτροπή, δηλαδή με μείωση 5%. Ε, τότε τι αλλάζει σε σχέση με το γενικό στόχο. Γιατί μία καταπερίπτωση προσέγγιση θα αλλάξει τα πράγματα. Τι διαφορά υπάρχει, αν ο στόχος είναι ο ίδιος. Και αν εκτιμάτε ότι μπορείτε να τον πετύχετε, τότε τι αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Εγώ δεν το κατάλαβα με αυτά που μας απαντήσατε. Ωραία, ποιος θα απαντήσει για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ο συνάδελφος. Μπορώ να του δώσω το λόγο, παρακαλώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Ντεπρές. Πρέπει να διευκρινιστεί κάπως εδώ το πράγμα. Στο έγγραφο το οποίο σας υποβάλαμε, οι οργανισμοί δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση της επιπλέον μείωσης 5% στον προπολογισμό σε σχέση με το 5% που ζητάτε από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μάλιστα με την προσέγγιση που ζητάτε. Δηλαδή, ένα κονδύλι για, όλες, για όλους τους οργανισμούς, τους αποκεντρωμένους και από την άλλη μεριά να ζητάμε από αυτές οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμα τον κανονικό ρυθμό εργασιών τους να ζητάμε μια παραπάνω προσπάθεια, αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και αυτό το λέμε και σε ένα άλλο έγγραφο. Γιατί το πρώτο είναι ότι το τι θα γίνει στη συνέχεια είναι λιγάκι ασαφές. Έπειτα, οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένου τομεί. Και όταν αναφέρθηκε στο ρόλο των επιτροπών, μεταφορών κτλ., μην ξεχνάμε το εξή. Ένας αποκεντρωμένος οργανισμός μία κοινή επιχείρηση μπορεί με συνεργασία να φροντίσει να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά ήδη είναι δύσκολο όταν είναι όλοι μαζί οργανισμοί. Στην καταπερίπτωση προσέγγιση σημαίνει ότι θα εξετάσουμε την περίπτωση του κάθε οργανισμού, αλλά θα λάβουμε υπόψη μας και την γενικότερη πολιτική που εφαρμόζεται. Και το άλλο είναι βέβαια λεπτομέρεια. Δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε τη συνοχή ανάμεσα στο γενικό κανόνα και μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε επικεφαλή στο Συμβούλιο. Έτσι. Τα κράτη-μέλη όμως δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους για την μείωση των καθηκόντων, για παράδειγμα, των οργανισμών. Συνεπώς, οι οργανισμοί δεν συμφωνούν με την επιπλέον προσπάθεια 5% που τους ζητάτε έτσι όπως προτείνεται. Η πρότασή μας είναι λοιπόν η προσέγγιση να είναι κατά περίπτωση, οπότε κατά περίπτωση και κατά πολιτικό τομέα να εξετάσουμε την πρόταση που γίνεται. Πολλοί από εσά είπατε να βάλουμε μαζί οργανισμούς ανά κατηγορία καθηκόντων. Εντάξει και το 2009 έγινε μία μελέτη που ζήτησε η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και εκεί διευκρινίστηκαν πολλά πράγματα. Η γενική μας θέση λοιπόν είναι δεν συμφωνούμε με την οριζόντια προσέγγιση για μία κατηγορία οργανισμών γιατί θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολιτικές, οι δραστηριότητες, είτε πρόκειται για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Δεν θέλουμε ένα κανόνα που να εφαρμόζεται σε όλους. Πρόεδρος αν υπάρχουν τρει με τέσσερι οργανισμοί που ασχολούνται με μια πολιτική, τι λέτε, λέτε ότι μπορούμε να βάλουμε μαζί αυτου του οργανισμου και ότι σε αυτή την περίπτωση κάποιοι μπορεί να κάνουν μια προσπάθεια 10% μείωση και κάποια άλλη λιγότερη. Κύριε Ντεπρέ, συγγνώμη λοιπόν, ή εγώ δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω, πάντως εδώ πέρα λέει ότι η προσέγγιση παντω εδω περα λεει οτι περίπτωση θα επιτρέψει να πετύχουμε το στόχο τη μείωση 5% σε κάθε όργανο. Εδώ δεν μιλάμε για ομαδοποίηση, δεν μιλάμε για κλάστερ, μιλάμε για κάθε οργανισμό. Το κείμενο θα τροποποιηθεί. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι λέει το κείμενο που έχω μπροστά μου. Απάντησε. Ναι, καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια 5% και θα την κάνουμε. Τα επιπλέον 5% που ζητάτε να κάνουν προσπάθεια μείωσης οι οργανισμοί, αυτό είναι με το οποίο δεν συμφωνούμε. Κάποτε είχαμε πει να παγώσει ο αριθμός και να μην υπάρξουν νέοι οργανισμοί. Αλλά δεν ήταν αυτό εφικτό. Έτσι κι αλλιώ η πιστοποίηση ενό τρένου υψηλής ταχύτητα ή ενό αεροπλάνου κτλ. δεν πρόκειται να μειωθούν. Το 5% λοιπόν ναι, θα το κάνουμε και εμείς όπως και όλα τα όργανα. Τα επιπλέον 5% είναι που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Δεν με έχετε πείσει γιατί στο κείμενο λέει ότι η πρότασή σας έχει σαν στόχο εναλλακτική λύση αντί για το redeployment pool. Δηλαδή ότι δέχεστε τα 5% αλλά θα τα πετύχετε με διαφορετικό τρόπο αντί να μπαίνει όλοι οι οργανισμοί μαζί να και δημιουργηθεί αυτό το pool προσωπικού που λέγαμε. Θα συνεχίσουμε. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο κύριε Ντεπρέ αν αυτό είναι απαραίτητο. Ε, Ούτω ή άλλω για τους οργανισμού και για τις θέσεις εγώ κατάλαβα πως ε, η εβδομάδα εργασία έχει περάσει από τις 7 ώρε στις 40. Μάλιστα. Χωρί να αλλάξουν οι μισθοί. Άστα, συνεχίζουμε. Συνεχίστε μάλλον. Τελευταίο σχόλιο, ναι. Έχει, έχει αυξηθεί, ναι. Τελευταίως, δύο μιλητές έχω να απαντήσω. Το κύριο Ετσενίκουε. Και πάλι έχουμε εκεί το θέμα της ομαδοποίησης των οργανισμών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για ομαδοποίηση. Μιλήσατε για την δικαιοσύνη, εσωτερικά ασφάλεια. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία επί της ουσίας, αλλά και για τα διοικητικά θέματα ανάμεσα στους οργανισμούς ε, ε, δικαιοσύνης εσωτερικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι μέσα στη, σε αυτή την ομάδα. Ε, Όπω είπε και ο Πρόεδρος, θα πρέπει να εξεταστούν άλλες μορφές ομαδοποίησης. Επίσης ρωτήσατε αν υπάρχει πλεόνασμα στους οργανισμούς. Όταν ξεκινά μια τέτοια διαδικασία, βλέπει κανείς τους οργανισμούς και εξετάζει πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων. Όχι ότι δεν έχουμε γενική εικόνα για τις 41 οργανισμούς ή όργανα, αλλά Μπορούμε πάντοτε να τα πάμε καλύτερα. Ναι, μπορούμε να εισάγουμε νέες τεχνολογίες για να εξοικονομήσουμε. Είμαστε λοιπόν επιποδός πολέμου για να προχωρήσουμε. Ε, αλλά χρειάζεται να ενισχυθεί ο διάλογος. Τελευταίος ο μιλητής, ε, ο κύριος Κόλμελ, μίλησε για λειτουργική ανάλυση των οργανισμών και το ρόλο που παίζουν στο συγκεκριμένο κάθε φορά τομέα. Και πάλι αυτό παραπέμπει στην περιπτωσιολογική ανάλυση. Εμεί θέλουμε να δούμε ακριβώς τι αναμένουμε από τους οργανισμούς. Έτσι, νομίζω εγώ απέντησα σε όλες τις ερωτήσεις που έχω εδώ στο δικό μου κατάλογο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Διευθυντή της ΓΙΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Προπολογισμού της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω απαντώντας στις ερωτήσεις που υποβάλατε εσείς, ο κύριος Κόλμελ, αλλά και άλλοι βουλευτές όσον αφορά την προσέγγιση, πώς δηλαδή θεσπίζουμε ή επεκτείνουμε τα καθήκοντα ή τον περίμετρο δράσης ενός οργανισμού. Πάντοτε περνάμε μέσα από μια νομοθετική διαδικασία όπου η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού ή την επέκταση των καθηκόντων, την αύξηση των καθηκόντων ενός υφιστάμενου οργανισμού. Αυτό είναι συνοδευόμενο από μια τελογική έκθεση, αλλά και από ένα ε, δημοσιονομικό δελτίο που ε, παρουσιάζει την αξιολόγηση, την εκτίμηση τη δημοσιονομική, που θα πρέπει να υπάρξει αύξηση κτλ. Εξαρτάται βέβαια από το κάθε οργανισμό κάθε φορά. Άρα λοιπόν στη φάση της δημιουργίας ή της επέκτασης των καθηκόντων κάποιου οργανισμού γίνεται εξέταση του θέματος και κρίση ε, όσον αφορά την πολιτική σκοπιμότητα και τη δημοσιονομική σκοπιμότητα όλων αυτών. Και εκεί υποχρεούμεθα, αφόσον ληφθεί απόφαση, να φτιάξουμε ε, τον οργανισμό ή να επεκτείνουμε, να διευρύνουμε τα καθήκοντα και εκεί επί τη βάση αυτών των εκτιμήσεων ε, η Κομισιόν αξιολογεί τις ανάγκες μέχρι το 2020 και αυτό το κάναμε αναπερίπτωση, δεν βάλαμε όλους τους οργανισμούς στο ίδιο καλάθι και δεν χρησιμοποιήσαμε ενιαίο τρόπο υπολογισμού και εκτίμησης. Αυτό όμως πρέπει να συνδυαστεί και να συμφιλειωθεί με τους κεντρικούς στόχους, το top-down, που είναι η επίτευξη της μείωσης 5% στο προσωπικό όλων των οργανισμών και ιδρυμάτων της Ένωσης για 5 χρόνια, μέσα σε 5 χρόνια. Η αναπερίπτωση λοιπόν ανάλυση δεν δίνει ως φυσιολογικό αποτέλεσμα μια μείωση 5%. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Εάν δούμε τα αιτήματα του συνόλου των αποκεντρωμένων οργανισμών για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015, το σύνολο μας δίνει 209 θέσεις επιπλέον. Αυτό σημαίνει 3,3% αύξηση και όχι 5% μείωση, ούτε καν ε, μείον 1%. θέλουμε να δώσουμε στους οργανισμούς τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σωστά, αλλά ταυτόχρονα τις ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν τις προσπάθειες εξορθολογισμού και αποτελεσματικότητας που ζητούμε από όλους. Έπειτα. αποκεντρωμένοι οργανισμοί και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Έχουμε ας πούμε τις συμπράξεις πρωτοβουλίας που είναι είτε συμπράξεις είτε υπό την αιγίδα του προγράμματος Horizon 2020, δηλαδή ε, το πρόγραμμα για την έρευνα. Και εκεί προσπαθούμε να ελκύσουμε προδιωτική συμμετοχή, αλλά και συμμετοχή των κρατών μελών για ορισμένα ερευνητικά προγράμματα και προσπαθούμε δηλαδή εκεί να συνδυάσουμε διάφορους πόρους χρηματοδότησης για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο οποίος λειτουργεί ως καταλητής για τις προσπάθειες που προέρχονται από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα της Ένωσης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μηχανισμοί που διαφέρουν κάπως σε δημοσιονομικό επίπεδο, ακόμα και αν σε διοικητικό επίπεδο υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά δεν είναι το ίδιο όπως μια υπηρεσία που έχει ε, κοινά καθήκοντα σε όλη την Ένωση και όπου συχνά πρέπει να συνδυαστούν αρμοδιότητες που ήταν διασκορπισμένες σε εθνικό επίπεδο για τις συμπράξεις τεχνολογικές ε, δεν ε, ισχύουν τα ίδια. Στη συνέχεια, ο κύριος Γκάιερ έθεσε το θέμα των εξωτερικών ελεγκτών για τους οργανισμούς και αν προβλέπετε κάτι ε, για να μπορούν οι οργανισμοί να έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Εμείς θέτουμε στη διάθεση των οργανισμών τους καταλόγους των, εξω... των ε, συγκεκριμένων ειδικών ελεγκτών που χρησιμοποιεί και η Κομισιόν και μετά ο κάθε οργανισμός ε, μπορεί να προβεί στην ε, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάλογα με το πώς διοργανώνει κάθε φορά τους διαγωνισμούς του. Να κοιτάξω αν έχουμε εδώ κάποιο άλλο στοιχείο. Ναι. Το πλαίσιο εντό του οποίου λοιπόν υπέβαλε την πρότασή της η Κομισιόν είναι ένα πλαίσιο με σταθερή πολιτική, δηλαδή με τις ε, ε, υφιστάμενους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των όσων δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Και ακριβώ εντό όλων αυτών επιδιώκεται το στόχο του 5%. Τώρα, για νέους οργανισμούς που προστίθεται, που φτάνουν στη συνέχεια, όπως είναι το Συμβούλιο Εξυγίασης για τις Τράπεζες, η Κομισιόν δεν ζητά να το λάβουμε υπόψη αυτό και να κάνουμε την αντίστοιχη εξοικονόμηση αλλού. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο πολιτικής που εισήχθη έκτοτε και το οποίο θα πρέπει χωριστά να εξεταστεί επί τη βάση νομοθετικής πρότασης που έχει υποβληθεί συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιονομικών επιπτώσεων, οικονομικών επιπτώσεων. Εάν κάτι ξέχασα, ζητώ συγγνώμη και είμαι έτοιμος, με στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτές οι διευκρινήσεις ε, ίσως να προκάλεσαν και άλλα σχόλια. Κύριε Ντεπρέ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ένα κομμάτι μιας ε, έμεσης ερώτησης, στην οποία δεν έλαβα απάντηση. Η μείωση του 5% που ζητάει η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που χρηματοδοτούνται από τους ίδιους πόρους των ε, οργανισμών. Διότι μπορώ να κατανοήσω ότι θα ληφθούν υπόψη όλα όσα επιβαραίνουν τον προπολογισμό. Γιατί ναι, εκεί όντω πρόκειται για περιορισμό των θέσεων που επιδοτούνται από τον, από τον προπολογισμό. Αλλά αν υπάρχουν θέσει στι οργανισμού που χρηματοδοτούνται από εξωτερικού πόρου, η Κομισιόν αυτό το λαμβάνει υπόψη ή όχι. Δηλαδή, εξαιρεί αυτέ τι θέσει από τη μείωση του 5%. Ναι, κύριε Πρέσα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προσέγγιση της Κομισιόν όλες οι θέσεις έχουν ληφθεί υπόψη. Και αυτό διότι από τη μια πλευρά η διαθεσμική, διοργανική συμφωνία δεν προβαίνει σε διάκριση ανάμεσα στο είδος της χρηματοδότησης των οργανισμών και δεύτερον θα έλεγα διότι ούτως ή άλλως η προσπάθεια ε, επίτευξης ε, ε, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και εξοικονομήσεων δεν έχει σχέση με το αν είναι χρηματοδοτούμενες οι θέσεις από τον προπολογισμό ή από τέλη τα οποία επιβάλλονται στον τομέα κάθε φορά. Όσον αφορά λοιπόν τον οικονομικό εξορθολογισμό, θα πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο αποδοτικότητος ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης. Η προσπάθεια λοιπόν κατανέμεται στο σύνολο των οργανισμών και στο σύνολο των θέσεων. Θα έλεγα επίσης ότι αναφερούσαμε τις θέσεις που χρηματοδοτούνται από τα τέλη που καταβάλουν οι κλάδοι καθορά. Θα, θα έλεγε κανείς ότι το σύνολο στο οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε για να ενισχύσουμε κάποιους οργανισμούς που πρέπει ακόμα να διευρυνθούν, θα σήμαινε ότι θα είναι ακόμα πιο μικρό αυτό το σύνολο και ορισμένοι οργανισμοί θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα περισσότερο από το 10% για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Ο κύριος Μάνκα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι οι οργανισμοί λένε ότι εάν μειώσουν κατά 5% μπορεί αυτό να μην αποβεί βάρος τους, όμως σε άλλους οργανισμούς η περικοπή αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις δαπάνες ορισμένων οργανισμών, αυτό χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να έχουμε πρώτα μια ξεκάθαρη εικόνα πού οι περικοπές αυτές είναι δυνατές και πού όχι. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει εξωτερικός έλεγχος θα είναι σκόπιμο να γίνει αυτός υπό την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να προβλεφθούν ενδεχομένω μέτρα λιτότητα σε έναν οργανισμό, ή περικοπές. Μπορεί ωστόσο να γίνει αυτό και στη βάση ενός κλάστερ, μιας ομάδας οργανισμών. Μπορούν να επιτευχθούν ίσως και διαφορετικά μεγέθη περικοπών ανά οργανισμό. Η προσέγγιση λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτική. Ποιο θέλει να απαντήσει, ρωτά ο πρόεδρο. Κύριε Κερούμ, εσεί κύριε Πρέσα. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αξιολόγηση του συνόλου των οργανισμών βεβαίως ως αίτημα είναι θεμητό. Βέβαια είναι ένα έργο μεγάλης εκτάσεως. Διορωτώ εάν μέσα στα πλαίσια των εργασιών της διαθεσμικής ομάδας θα πρέπει ενδεχομένως να μελετηθεί και αυτό για να υπάρξουν και κάποια στοιχεία ορθολογισμού. Για την ώρα πάντως αξιολόγηση του είδους αυτού δεν προβλέπεται. Ευχαριστώ. Ο Monsieur Κερούν. Για την ερώτηση αυτή και για να υπάρχει διαφάνεια Έφερα το παράδειγμα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έγινε αξιολόγηση των εργασιών του προδιετίας και σε τακτά διαστήματα κάθε 4-5 χρόνια θα ξαναγίνει. Γιατί τότε έχει κανεί αυτό το feedback από ένα σοβαρό εξωτερικό οργανισμό για το πώς γίνεται πώ λειτουργεί ο οργανισμό. και βέβαια και προ όφελο των stakeholder. Ένα από τα προβλήματα βέβαια που σημειώνονται εδώ με αυτέ τι εξωτερικέ αξιολογήσει, είναι ότι προσθέτουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή λένε τελικά καλά τα πάει ο οργανισμός αλλά θα θέλαμε να δούμε και τα εξής 1, 2, 3, 4, 5 κάνουν συστάσεις έξτρα δηλαδή. Ωστόσο αυτό τροφοδοτεί τη συζήτηση βέβαια. Σωστό είναι. Αν με επιτρέπετε τώρα να παρακαλέσω την διεύθυνση του Οργανισμού Ναρκωτικών Φαρμάκων διορθώνει ο Ε, μπορεί να σας εξηγήσει περισσότερο τη δική τους περίπτωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας μιλήσω για το δικό μου οργανισμό που θα σας δείξει πόσο διαφορετική είναι οργανισμική και γιατί χρειαζόμαστε ξεχωριστή εκτίμηση. Είμαι επικεφαλής του οργανισμού εδώ και πολλά χρόνια και πρόκειται τελικά όντως για τα ναρκωτικά και τοξικομανία και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης δραστηριοποιούμεθα. Και σημαντικό να σας πω σε εσάς εδώ ότι είμαστε μεταξύ των τριών κορυφαίων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού μας. 97% των πληρωμών μας. Πραγματικά έξοχο, ε, εξέχον έργο. Πρόκειται για οργανισμό της δεύτερης γενιάς με 20 ετή ηλικία και έχουμε ως σκοπό να αναλύουμε όλες τις πτυχές των παράνομων ναρκωτικών. Και βεβαίως εκτός από τα καθήκοντα αυτά που ασφαλώς δεν έχουν μειωθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να συζητούμε και τις νομικές πτυχές των νέων ψυχοτρόπων φαρμάκων. Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ βέβαια κάνουμε λοιπόν αξιολογήσεις κινδύνου με πολλές μελέτες με την επιστημονική μας επιτροπή που απαρτίζεται από 16 πανεπιστημιακούς καθηγητές και αυτά τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι το πιο δυναμικό τμήμα των, της λειτουργίας του οργανισμού μας. Έχουμε στο ραντάρ μας τώρα 400 ουσίες που παρακολουθούμε καθημερινά. Από το 1997, 75% των ουσιών εντοπίστηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο βαρύ είναι το έργο μας. Έχουμε σταθερό προπολογισμό από το 2010. Έχουμε καταφύγει τον πληθωρισμό και τα πάντα. Έχουμε αφομοιώσει τον πληθωρισμό, δεν έχουμε ε, ζητήσει ποτέ. Το μόνο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι να ακολουθούμε την πρόταση της Κομισιόν. Όμως πέρσι η Κομισιόν πρότεινε 5% περικοπή. Εμείς έχουμε και το Home Affairs Cluster, έχουν γίνει βεβαίως περικοπές. Έχουν γίνει αλλού αυξήσει που σίγουρα ήταν δικαιολογημένες και σε εμά ζητούνται περικοπές. Εν τέλει, στην συνολομέλειά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε την ε, περικοπή αυτή και ενέκρινε να επαναληφθεί για το 2014 ο προπολογισμό του 2013. Τελικά όμως στη συνδιαλλαγή κατέπεσε η θέση αυτή και έγινε η μείωση του 5%. Τώρα η Κομισιόν ζητεί να δεχθούμε τον προπολογισμό ξανά το 2014, δηλαδή, δηλαδή τη μείωση του 5%. Δεν ξέρω πώ θα αντεπεξέλθω στι νομικέ μου υποχρεώσει και θα εξασφαλίσω την ποιότητα του έργου μα που έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ νομίζω ότι πραγματικά χρειαζόμαστε ισότιμη μεταχείριση κάποια στιγμή και νομίζω ότι αυτή η περικοπή του περσινού χρόνου πρέπει να διορθωθεί. Όπω ζήτησε και η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συσκηνοβουλίου πέρσι τον Οκτώβριο μιλώ για ένα ειδικό δυναμικό τομέα με ειδική νομική βάση για τα νέα ψυχοτρόπα φάρμακα. Εκεί έχω πάρει όποιους πόρους βρήκα από αλλούς και τους έχω ρίξει εκεί. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Ο οργανισμός έχει φτάσει και ξεπεράσει τα όρια του. Ευχαριστώ. Στο έγγραφο σχετικά με τον οργανισμό σας βλέπω ότι για το προϋπολογισμό του 2014 είχατε 15 εκατομμύρια περίπου, για το 2015 έχετε πάλι 14 εκατομμύρια και λίγο λιγότερο. Βλέπω και other income, άλλα έσοδα, που πάνω από ένα εκατομμύριο φτάνουν τώρα σε 65.000. Πώς έγινε αυτό? Τα άλλα έσοδα είναι από ελέγχους, είναι τεχνική ενίσχυση σε χώρες και σε χώρες της ε, πολιτικής γειτονίας. Δεν έχει καμία, κανένα ιδιαίτερο νόημα για τον οργανισμό μας. Και το υπόλοιπο μέρος είναι 400.000 περίπου συμβολή της Νορβηγίας στον οργανισμό, που συναποτελεί ένα ποσοστό του προπολογισμού μας. Μερσίλιο, Πρόεδρος. Άλλες ερωτήσεις δεν έχουμε, άλλα σχόλια ούτε. Οι εκπρόσωποι των οργανισμών έχουν... Α, εσείς κύριε. Χωσέ Πενέρο του Οργανισμού Ασφάλειας των Εναέριων Μεταφορών. Για το δημοσιονομικό δελτίο νομίζω θέλω να σας μιλήσω, όπως και για την ΕΑΣΑ. Έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από τα 2 τρίτα, 80% στην ουσία, από τέλη που πληρώνει ο κλάδος. Αυτό δεν μπορούμε εμείς βέβαια να το επηρεάσουμε. Πρέπει να υποστηρίξουμε την βιομηχανία εναέριων μεταφόρων. Γιατί αυτή είναι βεβαίως η πρώτη στη εντολή μας είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας στην αέριες κυκλοφορές. Αλλά έχουμε και ειδική εντολή να υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία για να γίνει πιο ανταγωνιστική, να εξασφαλίσουμε εξοικονομήσεις υπέρ τους, να προωθήσουμε την ενιαία αγορά που ήδη έχουμε δημιουργήσει και αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις υπέρ της βιομηχανίας και να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική προς τα έξω. 80% λοιπόν το, του προπολογισμού μας χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία. Δεν έχει καμιά σχέση με τον κοινοτικό προπολογισμό. Και θα πρέπει να το σκεφτείτε αν όντω πρέπει να επιβάλλετε την περικοπή του 5% σε αυτό το τμήμα του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτές τις ευκρινήσεις. Θέλει κανεί άλλο το λόγο? Όχι. Ίσως μια ερώτηση για τον κύριο Πρέσα από τον αγγραφό του. Θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι για την κληρονομιά της κάθε μιας από, αυτές, από αυτούς τους οργανισμούς, τα περιουσιακά στοιχεία, αν υπάρχει κάτι που θα ήταν ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας. Mm. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ερώτηση αυτή γιατί μου επιτρέπει να κάνω και λίγο διαφήμιση για τα έγγραφά μας. Να, αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο επικεντρώνεται στους οργανισμούς. Είναι ένα έγγραφο εργασίας που συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού. Είναι 600 σελίδες και υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον καθένα από τους οργανισμούς αλλά και στο σύνολό τους για την ε, χρήση για πιο διοικητικές και δημοσιονομικές πτυχές επίσης. Η ερώτησή σας λοιπόν είναι κατά πόσο υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Όταν ετοιμάζουμε το σχέδιο προϋπολογισμού, λαμβάνουμε υπόψη την ε, χρήση της χρονιάς που πέρασε. Και αν υπάρχει πλεόνασμα, αν υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στις δαπάνες και τα έσοδα, τότε λαμβάνεται υπόψη αυτό για να υπολογιστούν οι επιδοτήσεις, η προκοδότηση για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή το πλεόνασμα αυτό ανακυκλώνεται στον ίδιο οργανισμό. Είναι ένα έσοδο το οποίο λαμβάνεται υπόψη ως τέτοιο. Και άρα έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε πιο σωστά τις πιστώσεις που θα δώσουμε και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό τα ποσά αυτά να εκφράζονται στον προπολογισμό πολύ συγκεκριμένα. Καμιά φορά αν υπάρχει πάνω από 5% του προπολογισμού πλεόνασμα, τότε εισάγουμε και ένα σύστημα προστίμου, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν παγώνουμε μεν τις πιστώσεις, στη χρηματοδότηση, αλλά μάλλον παγώνουμε τις πιστώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αντικίνητρο, άμα θέλετε, ο οργανισμός, ο κάθε οργανισμός, ε, για να κρατήσει πλώνασμα. Τώρα, σε περίπτωση αυτοχρηματοδότησης, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, όπου μαζεύτηκαν ε, χρήματα, κονδύλια όλα αυτά τα χρόνια, και μετά από συζητήσεις αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά σε προγράμματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Η δημιουργία πάντως ενός πλονάσματος που να συσσωρεύεται χρόνο το χρόνο είναι κάτι που πρέπει να δούμε σαν ανομαλία. Γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος να συσσωρεύονται πλεονάσματα, οι οργανισμοί χρηματοδοτούνται για να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες ε, στο κόσμο, στη βιομηχανία, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οπότε ο δημοσιονομικός υπολογισμός πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει συσσόρευση, περιττή συσσόρευση πλεονάσματος σε κάποιους οργανισμούς. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Καταλαβαίνω την απάντησή σας. Όμως, Υποθέτω ότι έχουν λογιστικά ε, βιβλία οι οργανισμοί αυτοί και εκεί αναφέρεται το ενεργητικό, το παθητικό κάθε φορά. Έτσι δεν είναι. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε και εμείς την εικόνα αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Μερικές φορές υπάρχουν εκπλήξεις, ξέρετε. για το τι μπαίνει στο αποθεματικό, για παράδειγμα. Θα ήταν μια παραπάνω πληροφορία για μας, βλέπετε. Καλώς, αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τότε σας ευχαριστώ όλους την αντιπροσωπεία πρώτα απ' όλα των οργανισμών, την Τρόικα που ήρθε να μας παρουσιάσει την κατάσταση των οργανισμών, τις δυσκολίες τους, την ανάγκη για μείωση του διοικητικού κόστου, του προσωπικού, παρόλο που μερικές φορές να λαμβάνουν νέα καθήκοντα. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Πάντα είναι εύκολο να λέμε ότι κόβουμε παντού το ίδιο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προσέξουμε όλους ιδιαίτερως την κάθε μία χωριστά από αυτέ τι υπηρεσίε, από αυτού του οργανισμού. Να του δούμε χωριστά έναν ένα για το καθένα έχει ιδιαιτερότητε. Μπορούμε ίσω να φτιάξουμε κάποιε ομάδε για να δούμε τι κοινά έχουν μεταξύ του να τις ε, ταξινομήσουμε, να ταξινομήσουμε τους οργανισμούς αυτούς μαζί μερικές φορές, αν έχουν ε, παρόμοια καθήκοντα. Μπορεί να βοηθούσε αυτό. Οπότε, εσείς που είστε υπεύθυνοι των οργανισμών, αλλά και εσείς από την Επιτροπή Προϋπολογισμών όλοι να είσαστε πολύ προσεκτικοί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μέχρι τώρα προσπάθειές σας για να μας δώσετε εγγύησει για καλή διαχείριση. Εγγύησει για να πετύχει η μείωση αυτή των δαπανών. Τώρα ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των ιδιών πόρων που θα ήταν πηγή χρηματοδότησης αυτή για διάφορους οργανισμούς ενώ έχουν θεσμικό βέβαια έργο και στόχος τους είναι η ρύθμιση των τραπεζών για να αποφεύγονται νέοι συστημικοί κίνδυνοι. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, αυτοί οι οργανισμοί που βέβαια πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι, παρόλα αυτά βάσει συγκεκριμένων νομικών διατάξεων που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο θα μπορούσαν να βρούνε και άλλους πόρους και άλλα έσοδα για να υπάρχει ισορροπία στον προπολογισμό τους. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λοιπόν που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Θα τα ξαναπούμε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Υπάρχει τίποτα άλλο? Όχι. Συνεπώς, σας εύχομαι καλές διακοπές σε όλους. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί από τις 3 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι σε συνεδρίαση. Οι δημοσιονομικές διαιτησίες, όπως καταλαβαίνετε, θα μας κινητοποιήσουν πάρα πολύ το φθινόπωρο για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους απλήρωτους λογαριασμούς που έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλές διακοπές και σας ευχαριστώ. άλλη συνεδρίαση.